Έχει παρέλθει το ακαδημαϊκό τέταρτο, αγαπητοί συνάδελφοι. Οπότε μετά από αυτό το ακαδημαϊκό τέταρτο θα περάσουμε και εμείς σε μια συζήτηση πολύ σημαντική, σφαιρική. Ε, δεν ξεχνούμε βέβαια ότι σήμερα είναι Δευτέρα και πολύ έρχονται τώρα στις Βρυξέλλες, πολλοί ευρωβουλευτές. Και μάλιστα είχαμε και ένα τραγούδι στην Πολωνία, δεν μ' αρέσει η Δευτέρα, δεν ξέρω γιατί. Τσάκαρο Δευτέρα που λέμε. Ε, ας δούμε την ημερήσια διάταξη και να την εγκρίνουμε. Και να δούμε κάποια διαδικαστικά. Καταρχήν μεταδίδεται στο διαδίκτυο η απογευματινή μας συνεδρίαση. Έχουμε διερμήνει από και προς 20 γλώσσες, με εξαίρεση τσεχικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και γοητελικά, κελτικά. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 23ης και 24ης Ιανουαρίου, 29ης Ιανουαρίου και 7ης Φεβρουαρίου. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις, μέχρι το τέλος της συνεδρίας θα θεωρηθούν συγκεκριμένα τα Οπότε περνάμε στο ένα και μοναδικό κυρίως θέμα, ουσιαστικό ζήτημα της απογευματινής μας ημερήσης διάταξης, που είναι η ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Κατρίν Γκελάν Λανέλ, υποψήφια και τη θέση της Γενικής Διευθύντριας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων και μάλιστα η συνεδρία αυτή γίνεται από κοινό με την Επιτροπή Ανάπτυξης, την ΤΕΒΕ, και θα ήθελα να καλωσορίσω ε, την ε, Πρόεδρο και θα της δώσω όσον από το λόγο της Συμπροέδρου. Αυτά είναι ήδη εισαγωγή. Να καλωσορίσω και πάλι θερμότατα την ε, καλεσμένη μας, την υψηλή μας καλεσμένη, την υποψήφια που σας είπα για τη θέση του Γενικού Διευθυντού ε, σε μια πολύ σημαντική οργάνωση παγκοσμίω γιατί αφορά τα τρόφιμα και τη γεωργία στον κόσμο. Θα έχουμε λοιπόν μια ανταλλαγή απόψεων. Πολύ συχνά έχουμε ανταλλαγές απόψεων με εκπροσώπους της ΦΑΟ, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, και χαιρόμαστε γιατί έχουμε ιδιαίτερα αγαστή συνεργασία. Η κυρία Κατρίν Γκελά είναι η πρώτη γυναίκα υποψήφια και μάλιστα κοινή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκλογή του Γενικού Διευθυντέ θα γίνει στην 41η διάσκεψη του ΦΑΟ τον Ιούνιο του 2019 και ο υποψήφιος ή η υποψήφια θα αναλάβουν ε, τα καθήκοντά τους την 1η Αυγούστου 2019. Μάλιστα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ε, υποψηφιότητα είναι 28 Φεβρουαρίου του 2019. Και μάλιστα η κυρία Γκελά είναι γεωπόνος, ε, έχει πολύ ψηλή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ασφάλεια ε, συστημάτων τροφίμων, αγροτική ανάπτυξη, ασφάλεια τροφίμων στη Γαλλία και στην Ευρώπη και έχει καταλάβει πολύ ψηλέ θέσει στο, Υπουργείο, στο Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν εκτελεστική διευθύντρια τη ε, Ευρωπαϊκή Αρχή, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων για 7 συνέχεια χρόνια και επίση ε, συμμετείχε σε πολλές ευρωπαϊκές και διεθνείς επιτροπές, συμπεριλαμβανομένων της Επιτροπής για το Κόντεξ Alimentarius και τις Γενικές Αρχές. Όπως γνωρίζετε, τα θέματα των τροφίμων και της γεωργίας ε, απασχολούν ε, συχνά και την Επιτροπή ΔΕΒΕ και ε, γι' αυτό έχουμε και κοινέ συνεδριάσεις Ε, για να εξετάσουμε είτε μονομένα προβλήματα χωρών ε, σε σχέση με τα τρόφιμα ή τη γεωργία ή παγκόσμια προβλήματα για τα θέματα αυτά. Οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκελέν, ε, στην συγγνώμη, στην πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, εγώ θα μιλήσω Ολλανδικά. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εκ μέρους της Επιτροπής ΔΕΒΕ Ε, χαίρομαι που μας δίνετε ευκαιρία να έχουμε μια κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Άγκρη και Ντέβε για να συζητήσουμε με την κυρία ε, Γκελέν Λανέλ. Η πρόεδρος της Επιτροπής ε, Ντέβε, η κυρία Λίντα Μαγκάβαν, δυστυχώς κολλείεται σήμερα και γι' αυτό την ε, αναπληρώνω εγώ. Χαίρομαι ιδιαίτερος για την ευκαιρία που μας δίνετε να ανταλλάξουμε απόψεις με την κυρία Γκέλα Λανέλ που θα μας πει πώς βλέπει το ρόλο του ΦΑΟ ε, σε σχέση με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όπως κλιματικές αλλαγές, το οικολογικό αποτύπωμα της γεωργίας και ούτω καθεξής. Είναι πολλές οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στην προσπάθεια να εξασφαλίσουμε επαρκή τρόφιμα για ολόκληρο τον πλανήτη. Και φυσικά η επάρκεια τροφίμων είναι ένα οξύ και φλέγον ζήτημα και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Γι' αυτό και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους οργανισμούς και τους φορείς των Ηνωμένων Εθνών είναι πολύ σημαντική. Μάλιστα για πρώτη φορά έχουμε κοινό ευρωπαϊκό υποψήφιο και μάλιστα γυναίκα υποψήφιο για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΦΑΟ. Ε, είναι πολύ πυρή η κυρία Γκελάν, πολύ εντυπωσιακό το βιογραφικό της και είναι σημαντικό να αναλάβει η Ευρώπη ηγετικό ρόλο στο ΦΑΟ προωθώντας τα ζητήματα των τροφίμων και της γεωργίας. Είναι σημαντική αυτή η θέση και η υποψηφιότητα της κυρίας Γκελάν λαμβάνει η χώρα σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, τη στιγμή προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια παγκόσμια επιστημιστική ασφάλεια. Και πρόσβαση των πάντων σε ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα. Ε, θορυβηθήκαμε ιδιαίτερως από τις τελευταίες μελέτες και εκθέσεις που δείχνουν ότι έχει 820 εκατομμύρια συνανθρώπων μας ε, υποσυτίζονται μονίμως και 151 εκατομμύρια παιδιά έχουν καχεκτική ανάπτυξη λόγω του υποσυντισμού. Δηλαδή η πείνα δυστυχώς δεν έχει καταπολεμηθεί επαρκώς. Οπότε εκτός από την, τον υποσυτισμό και την ασφάλεια τροφίμων έχουμε και μια τρίτη συνιστόσα στις, προσκλη, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε που είναι η αυξανόμενη παχυσαρκία παγκοσμίω που συμβαδίζει δυστυχώς με τον υποσυτισμό σε ορισμένες χώρες. Αυτές λοιπόν είναι αρκετά ανησυχητικέ τάσεις και μάλιστα εμείς ε, από το 1940 που είχαμε 80% πείνα, τώρα έχουμε φτάσει στο 4% και επιπλέον οι πιστώσεις ε, έχουν αυξηθεί αισθητά για το 2017. Οπότε, αν αναλάβετε την Γενική Διεύθυνση του ΦΑΟ, κυρία Γκέλα, θα πρωτοστατήσετε σε μια παγκόσμια προσπάθεια καταπολέμησης του υποσυτισμού και ε, υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τη μεγάλη σημασία που έχει η υλοποίηση αυτών των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Και με αυτή την άποψη με ενδιαφέρουν ε, τα σχέδιά σας και οι προτεραιότητες σας. Τι σκοπεύετε προκειμένου η ασφάλεια των τροφίμων να γίνει ύψη προτεραιότητα του ΦΑΟ και να πείσετε και με ποιο τρόπο θα πείσετε τα κράτη-μέλη να ειστεριστούν αυτό το στόχο. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω το λόγο κυρία Γκελάν Λανέλ και να σας παρακαλέσω να μην ξεπεράσετε το τέταρτο για να έχουμε το χρόνο για μια συζήτηση με τα μέλη των δύο επιτροπών. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων, κύριε Αντιπρόεδρε τη Επιτροπή Ανάπτυξη, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα καταρχά να σα ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σα που πήρατε την πρωτοβουλία για την ακρόαση αυτή. Και έχω την τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι εδώ ε, μεταξύ σα, μεταξύ των Ευρωβουλευτών, για να ανταλλάξω τι ε, απόψεις σε ό,τι αφορά τα θέματα επιστημικής ασφάλεια και ασφάλεια των τροφίμων και ξέρω πόσο πολύτιμέ και χρήσιμε είναι αυτές οι συνταλλαγέ απόψεων σήμερα, όπω ε, αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Είμαι ανάμεσά σα και σα παρουσιάζομαι ω υποψήφια από τη Γαλλία και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την, διεύθυνση, για την θέση τη Γενική Διευθυντρία ε, του ΦΑΟ. Το 2019 λοιπόν θα είναι σημαντική χρονιά για το ΦΑΟ σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή και το προσωπικό για όλους μας, γιατί θα εκλεγεί νέος γενικός διευθυντής. Όπως γνωρίζετε, η υποψηφιότητά μου υποβλήθηκε στη Γαλλία στις 17 Δεκεμβρίου και η υποψηφιότητα αυτή αποτελεί μια φιλόδοξη πρόκληση και γι' αυτό λοιπόν με την, με την υποστήριξη του Πρόεδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας του κ. Εμμανουέλη Μακρόν ε, την υποψηφιότητά μου πριν από την περίοδο Τη ε, ψηφιότητων. Του τελευταίου έξι μήνε λοιπόν ε, αφοσιώθηκα με ενθουσιασμό για να ξεκινήσει ένα διάλογο με τι κυβερνήσει και με του εμπλεκόμενε φορεί. Ε. Και προτίμασα λοιπόν τι προτεραιότητά μου και το σχέδιό μου για την ΦΑΟ. Και όταν ξε... ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου τον Ιούλιο, ξεκίνησε το διάλογο με περιφερειακές και διεθνεί οργανώσει, κυβερνήσει, τοπικέ κυβερνήσει. Αγρότε στον ακαδημαϊκό κόσμο και όλου του οικονομικού φορεί στην αλυσίδα τη των τροφίμων και με την κοινωνία των πολιτών με σκοπό να τροφοδοτήσω ακριβώ το έργο και τι προτεραιότητέ μου. Μόλι επέστρεψα από την Αντίζα Μπέμπα και από την Αίγυπτο και θα μεταβώ σύντομα στην περιοχή του Ειρηνικού και σκοπεύω επίση να επισκεφτώ την Λατινική Αμερική και την Ασία. Θα δράξω κάθε ευκαιρία να βρεθώ επί τόπου και να έχω άμεση ανταλλαγή με τους αγρότες, τους ε, ψαράδες και τις τοπικές κοινωνίες. Επίσης συμμετείχα και στη διαδικασία για τον διορισμό ενός ε, και μόνο υποψηφίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση που πλέον έχει ολοκληρωθεί. Και είμαι περήφανη που είμαι η υποψήφια πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη σε ό,τι αφορά την ε, εκλογή αυτή Διδαχόμενη από τα παθήματα του 2011 όπου δύο Ευρωπαϊκοί, είχαμε δύο υποψηφίου από την Ευρώπη και κανείς δεν εκλέχθηκε. Ξέρουμε ότι ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί στη διαδικασία ορισμού ενός και μόνο υποψηφίου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούμε τη σημασία τη διεθνού συνεργασία και τη πολυμέρεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη εκπροσωπούν το ίμιση των, της ε, επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Μία και μοναδική λοιπόν υποψηφιότητα αποτυπώνει τον ρόλο κλειδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΦΑΟ ως ενεργό μέλος για όλες τις δραστηριότητε. Επιπλέον, η ΦΑΟ είναι η μοναδική οργάνωση της Ευρωπαϊκής του, του ΟΗΕ που, είναι, που έχει πλήρως μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη από κοινού συμβάλλουν πάνω από 40% της χρηματοδότησης της ΦΑΟ σε ό,τι αφορά τις ε, υποχρεωτικές και τις εθελοντικές Είμαι υποψήφια από τη Γαλλία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι οι στόχοι μου και το έργο που έχω κατά νου είναι καθολικό και παγκόσμιο και θα ήθελα να συνενώσουν όλες τις χώρες μέλη τη ΦΑΟ. Και αυτό το project, αυτό το έργο θέλω να το χτίσω μαζί σας. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. είπατε, η πείνα είναι σε ανωδική τάση πάλι. 821 εκατομμύρια άτομα εξακολουθούν να υφίστανται πείνα. Ο αριθμός αυτός είναι ίδιος όπως και πριν από 10 χρόνια. 2 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, είναι υποζωτίζονται. 10% του πληθυσμού του κόσμου στις σε συνθήκες ακραίας και παράλληλα οι ΠΟΕ και η ΦΑΟ εξακολουθούν να, επι, να επιβεβαιώνουν ότι η επιδημία της παχυσαρκίας εξακολουθεί να αυξάνεται οι δημογραφικές εξελίξεις, οι αλλαγές στις δίαιτες, οι αλλαγές του κλίματος και η ανάγκη να αναδομηθούν τα οικοσυστήματά μας είναι όλα προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και η δυνατότητά μας να πετύχουμε τους βιώσιμους στόχους μέχρι το 2030 αποτελεί μια τεράστια πρόκληση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε όπως ενεργούσαμε ως τώρα. Λες και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη να αναλάβουμε δράση. Έχουμε λοιπόν λύσεις. Ναι, υπάρχουν λύσεις. Για να εφαρμοστούν λοιπόν αυτέ οι λύσει, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και των εμπλεκομένων φορέων. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη ΦΑΟ. Χρειαζόμαστε τη ΦΑΟ για να παρέχει ε, τη γνώση βάσει τεκμηρίων, βάσει επιστημονικών ε, στοιχείων και να παρέχει και λύσει. Χρειαζόμαστε επίση τη ΦΑΟ ω μια πλατφόρμα για διάλογο και συγκεκριμένη δράση για να τονωθεί η συνεργασία και οι συνεργαστικέ σχέσει. Χρειαζόμαστε τη ΦΑΟ ως κινητήρια μηχανή για την ανάπτυξη μέσω τεχνικής ε, συνεργασίας και αρρωγής και παροχή πολιτικής ε, συμβουλή τη κυβερνήση. Και σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα κάποιες από τις βασικές προκλήσεις που έχω για τη ΦΑΟ. Θα ήθελα καταρχά να εξασφαλίσουμε και να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι νέοι, όπω και όλε οι γυναίκε και οι άντρε που μέρα με τη μέρα είναι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία παραγωγή των τροφίμων αποτελούν το επίκεντρο τη δράση μα και των πολιτικών μα. Θα πρέπει λοιπόν μαζί του να συνεργαστούμε και μαζί του να μιλήσουμε. Θα ήθελα επίση να λάβουμε δράση προκειμένου η ασφάλεια τροφίμων, η γεωργία, τα συστήματα διατροφή, η αλληλεία και η δασοκομεία θα ξαναμπούν στο επίκεντρο τη πολιτική ατζέντα. Οι τομεί αυτή δεν είναι τομεί ε, του παρελθόντος. Είναι απαραίτητη και κρίσιμη για το μέλλον μας. Αυτή η τομή επίσης διδραματίζει σημαντικό ρόλο για να υπάρχει ασφαλής, υπάρχουν ασφαλή και τρεπτικά τρόφιμα για όλους. Επιπλέον υπάρχουν βασικές οικονομικές δραστηριότητες και ενέργειες για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης στην Ήπεθρο, οι οποίες είναι βασικές και για την αναγέννηση των οικοσυστημάτων μας και την προστασία του κλίματος. Και συνολικά αυτές οι λύσεις θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε και την ε, ατζέντα του ΟΗΕ για την ε, ειρήνη, την ευημερία, του πολίτες και του πλανήτη. Θα πρέπει να περιορίσουμε τις απώλειες ε, στην αλυσίδα διατροφής. Και επίσης θα πρέπει παράλληλα να προστατεύσουμε το κλίμα όπως και τους πολύτιμους φυσικούς μας πόρους όπως το νερό, τα εδάφη, τα δάση και τη βιοπικιλότητα. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η ΦΑΟ θα μας βοηθήσει να δραστηριοποιήσουμε κινητοποιήσουμε πιο πολλέ ε, δημόσιε και δυτικέ επενδύσει και πιο πολλέ καινοτομίε σε ό,τι αφορά τα συστήματα τροφίμων. Όπου και αν βρίσκονται οι κοινότητε στην Ήπεθρο, είτε είναι σε μικρά νησιά, είτε είναι σε περιοχέ που μαστίζονται από την ξηρασία και από την απερίμωση είτε βρίσκονται σε μια πολύ παραγωγική περιοχή όπου η ποιότητα του νερού θα πρέπει να αναδομηθεί σε μια περιοχή που πλήττεται από ζωνόσους ή από συστήματα φυτών θα ήθελα η ΦΑΟ σε κάθε περίπτωση να βοηθήσει κάθε χώρα να βοηθήσει τις ε, κυβερνήσεις ε, να βρει σωστές λύσεις. Αν θέλουμε να πετύχουμε, χρειαζόμαστε μια συλλογική ανταπόκριση. Καμία χώρα και κανένα φορέα δεν μπορεί να πετύχει μόνο του. Η ΦΑΟ είναι ο κοινό μα οίκο. Θα πρέπει μαζί να συνεργαστούμε και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μα. Όλε τι μορφέ συνεργασία. Συνεργασία νότο-νότο, μεταξύ νότου και βορρά. Και μια τριγωνική συνεργασία, μια και θα πρέπει να κινητοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη, το ταλέντο και τη γνώση που υπάρχουν παντού σε κάθε περιφέρεια του κόσμου. Η ΦΑΟ έχει ακόμα πολλά πετύχει, έχει πετύχει πολλά ως τώρα. Έχει σημαντικούς πόρους και από πλευρά ανθρώπινων πόρων και οικονομικών πόρων. Όμως πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα, να απτύξουμε εταιρικέ σχέσεις, συνεργασίες και ε, πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε ειδοποιώς διαφορά. Αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις, όμως θέλω να σας πω είμαι πεπισμένη ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και όπως ε, αυτά που καταφέρουμε τις τελευταίες πέντε δεκαετίες είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε τριπλασιάσει την παγκόσμια επιστημιστική παραγωγή. Ε, ο Παγκόσμιο πληθυσμό έχει αυξηθεί κατά 2,5 φορέ. Πρέπει όμω να συνεχίσουμε τι προσπάθειε μα, έτσι ώστε τα συστήματά μα για την παραγωγή τροφίμων να είναι πιο βιώσιμα, να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε καλύτερη απάντηση στι ανάγκε του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ΦΑΟ έχει συγκεντρώσει μοναδική γνώση και τεχνογνωσία, είναι σε θέση να βοηθήσει τι κυβερνήσει για να αναζητήσουν εφαρμόσιμε λύσει που θα μπορούν να καλύψουν τι ανάγκε και προτεραιότητέ του. Χρειαζόμαστε τη ΦΑΟ για να είναι πιο ευάλικτη, πιο διαφανής. Ε, ε, χρειαζόμαστε περισσότερους στόχους, προσιλωμένοι στο στόχο να είμαστε πιο καινοτόμοι και πιο αποτελεσματικοί. Η ΦΑΟ πρέπει να ενταχθεί πλήρως στο σύστημα των ΗΕ με ε, ουσιαστική συνεργασία με άλλους οργανισμούς των ΗΕ και κυρίως με το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα και το Διεθνές Ταμείο για την Γεωργική Ανάπτυξη, το αποκαλούμενο IFAD. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι η μετατροπή των επιστημιστικών συστημάτων είναι αναγκαιότητα. Τα συστήματα αυτά πρέπει να είναι περισσότερο προστατευτικά, αποτελεσματικά, χωρίς αποκλεισμούς, ε, να αντέχουν περισσότερο. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε ασφαλή τρόφιμα, διατροφικά ποιοτικά, ε, επίσης, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Για να μειώσουμε την πείνα και τον υποσυτισμό, πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε το σύστημά μας στις ανάγκες των πολιτών, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και ποσότητας. Έτσι ώστε οι πολίτες και οι κοινότητες ε, να μπορούν να ευημερούν στο χώρο τους και γι' αυτό οφείλουμε να βελτιώσουμε την ε, αξία αλυσίδας την αλυσίδα αξία. με συγχωρείτε. Ο βασικός μου στόχος είναι να υπάρχουν βιώσιμα τρόφιμα για όλους και είμαι ακράδαντα πεπισμένη ότι η ΦΑΟ μπορεί να μας βοηθήσει όλους για να επιτύχουμε. Η υποψηφιότητά μου αποτελεί την πρώτη υποψηφιότητα από τη Γαλλία προ την Γενική Διεύθυνση τη ΦΑΟ. Και θα πρέπει να σα πω ότι είναι και η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παρουσιάζει μία και μόνη υποψηφιότητα για τη θέση αυτή. Δεν είναι η πρώτη φορά που η γυναίκα είναι υποψήφιο με από την ίδρυση του ΦΑΟ στο 1945. Με την υποστήριξή σας, με την κινητοποίησή σας, την ενέργειά σας και την... Θέλω να είμαι η πρώτη γυναίκα, η πρώτη γυναίκα από την Ευρώπη στη διεύθυνση της ΦΑΟ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά κυρία Γκέλα. Παίρναμε τώρα στη συζήτηση με την Ομίγυρη και σε ερωτήσει των Ευρωβουλευτών. Ο κύριος Μποβέ ζήτησε πρώτος το λόγο. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ε, μία παρατήρηση επιτρέψτε μου πρώτα. Γιατί Όσοι δεν γνωρίζουν την ε, Κατρίν Γκέλα, την πρεσβύτερη, μπορώ να σου πω ότι για πολλά χρόνια είχαμε συνεργαστεί ε, με την κυρία Γκέλα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων και η πρόοδος που σημειώσαμε την επταετία ε, στην οποία ήταν πρόεδρος τη ΕΦΣΑ άλλαξε τον τρόπο λειτουργία αυτού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλεια Τροφίμων και ενίσχυσε τη διαφάνεια. Η κυρία Κελά ήταν η πρώτη που έβαλε κάποια τάξη και στα θέματα των μελετών και στην εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλεια Τροφίμων. Γιατί ε, ο οργανισμό αυτό ήταν πολύ συχνά πεδίο έντονων ε, εντάσεων και τριβών. Πάντως έγινε ένα σημάζεμα των εργασιών και η διαφάνεια χάρη στην κυρία Γκελά. Αυτή μια προκαταρκτική παρατήρηση. Η ομιλία ήταν εξαιρετική, αλλά δεν ε, αναφέρατε τίποτα για την επιστηστική κυριαρχία, δηλαδή το δικαίωμα των λαών ε, να έχουν μια επάρκεια, να εξασφαλίσουν τα τρόφιμα από την τοπική τους γεωργία. Μάλιστα εγώ το 1996 πήγα για πρώτη φορά στο ΦΑΟ και εκεί άκουσα για πρώτη φορά αυτό τον όρο της επιστηστικής κυριαρχίας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τις χώρες του Νότου κυρίως. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το θέμα, ε, πώς βλέπει το θέμα αυτό η μέλουσα διευθύντρια του, ΦΑΟ, του ΦΑΟ και μάλιστα είμαι θερμός υπέρμαχος αυτής της υποψηφιότητας, ο κύριος Κολομπιέ. Συγχαρητήρια, κυρία μου που είστε υποψήφια της Γαλλίας φυσικά και η μοναδική Ευρωπαία υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Διευθυντού του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα τρόφιμα και τη γεωργία. Θα έχετε απέναντι σας πολλούς υποψηφίους από πολλές και διάφορες χώρες, από πολλές υπήρους Γι' αυτό και σημειώνουμε την υποψηφιότητά σα και σα ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε να μα παρουσιάσετε το όραμά σα για μια γεωργία που θα σέβεται περισσότερο την υγεία των καταναλωτών, αλλά θα σέβεται περισσότερο και του γεωργού και την υγεία του. Είπατε ότι απέναντι στην παγκόσμια δημογραφική πρόκληση ε, θα ήταν δυνατόν να παράγουμε περισσότερα και καλύτερα. Και αυτή η πρόκληση είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν ε, πολλά θέματα που είναι σημαντικά για τη γεωργία μας και για την υπεθρό μας. Το θέμα της ε, επιστηστικής κυριαρχίας είναι πολύ σημαντικό. Και ε, η πρώτη μου απορία αφορά την ισχύουσα κοινή γεωργική πολιτική. Ποια είναι η θέση σας για τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ που αφορά κυρίως τις άμεσες ενισχύσεις που λαμβάνονται από ένα μικρό αριθμό γεωργών και κυρίως ε, μεγάλο γεωργών, μεγαλοκαλλιεργητών. Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2020 είναι αυτή τη στιγμή αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Εσείς πώς βλέπετε τη μείωση των γεωργικών κονδυλίων, τη συρρήκρωση του γεωργικού προϋπολογισμού που πρότεινε για το μέλλον της ΚΑΠ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης πώς βλέπετε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ελεύθερων Συναλλαγών και τη ε, διμερή διαπραγμάτευση ελεύθερων συναλλαγών με τον Καναδά, με τη ΣΕΤΑ ή συμφωνία με το Μερκοσούρ, τέτοιες διμερείς συμφωνίες θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Φυσικά η, τα πρότυπα α, οι ασφάλειες και υγιεινή τροφίμων στι στις χώρες αυτές είναι πολύ συχνά χαμηλότερα από τα δικά μας. Ενώ εμείς έχουμε ως έμβλημά μας την παραγωγή τροφίμων, υγιεινών και πολύ ποιοτικών. Σα ευχαριστώ και περιμένω τις απαντήσεις. Ο κύριο Ερντό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Ιρλάνδα, υποψήφια για την ε, θέση τη γενική Διεύθυνση τη ΦΑΟ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, το γεγονό ότι έχει καθεωρηθεί στις 7 ε, Ιουνίου η, η ημέρα της επιστησικής ασφάλειας. Η επιστημική ασφάλεια είναι κάτι το οποίο δεν θεωρούμε δεδομένο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό στην καθημερινή μας ζωή, γιατί χωρίς την επιστημική ασφάλεια υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και προφανώς ε, συνεκδοχικά και για την ε, οικονομία. Πρόσφατα είχαμε κάποια σκάνδαλα σε ό,τι αφορά τη σαλμονέλα ε, σε πουλερικά από την, ε, από την ε, Βραζιλία και ζητήματα με τα κινέζικα την ουσία μελιούς του Κίνα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποια είναι κατά τη γνώμη σας ε, η... ο ρόλος της ΦΑΟ σε τέτοια ζητήματα. Ε, κυρία Χόιμπος. Σας ευχαριστώ πολύ θέλω να σας πω το εξής. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που όσον αφορά αυτά τα οποία θέλετε να προάγετε, κυρίως, δηλαδή τους νέους, νομίζω ότι αν ρίξουμε μια ματιά στην Αφρική, θα δούμε ότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται μια προοπτική για το μέλλον. Χρειάζονται εργασία. Εσείς λοιπόν ε, στοχεύσατε κυρίως ε, στη βιωσιμότητα, στο να υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή αλλά και προστασία του κλίματος ε, Νομίζω όλα αυτά πολύ σωστά τα θέσατε. Μέχρι τώρα η ΦΑΟ είχε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο και στρατηγικά σωστό πρόγραμμα, κυρίως όταν πρόκειται για τη γεωργική οικολογία. Έχει, έχουμε μια συγκεκριμένη μέθοδο. Τώρα, κατά πόσο θα μπορέσουμε να τα επιτύχουμε όλα αυτά τα οποία μας αναφέρατε, αυτό θα φανεί βέβαια, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά που είπατε ε, συμβαδίζουν πολύ καλά και με την επισητιστική κυριαρχία που ανέφερε ο σε συνάδελφός μου. Γιατί ε, στην περίπτωση αυτή, ευθύ εξ αρχή λαμβάνουμε υπόψη μας την κοινωνική οικολογία. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εσείς ε, όσον αφορά την γεωργική οικολογία, τι ακριβώ προτίθεστε να κάνετε. Γιατί τώρα από ό,τι φαίνεται ε, θα επενδυθούν περισσότερα χρήματα από τη ΦΑΟ. Εσείς ε, θα συνεχίσετε να στείλετε υποστηρίζετε αυτή την άποψη. Και κάτι άλλο. Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού τη ΦΑΟ έχουμε συνάψει μια συμμαχία, τη συμμαχία κατά της πείνας. Βέβαια η συμμαχία αυτή είναι νεόκοπη, ε, τέτοιου είδους συμμαχία όμως δεν υπάρχει ακόμα στα εθνικά κοινοβούλια. Το φθινόπωρο έλαβε χώρα ένα μεγάλο συνέδριο στη Μαδρίτη και μετά η Ισπανική κυβέρνηση συνέστησε μια τέτοια συμμαχία για την αντιμετώπιση της πείνας. Μήπως έχετε και άλλες ιδέες για το πώς μπορούμε όλα αυτά να τα περάσουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια. Γιατί αν το κάνουμε αυτό θα έχουμε ένα πολύ καλό μοχλό για βελτίωση της συνεργασίας, κάτι το οποίο στην αρχή της ομιλίας σας εσείς παρουσιάσατε ως απολύτως απαραίτητο. Δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα όλα αυτά που μας είπατε να τα προάγουμε και σε κοινοβούλια κοινοβουλευτικό επίπεδο και μέσω των κοινοβουλίων και στις κυβερνήσεις. Ε, καλή τύχη σας εύχομαι, ελπίζω να διοριστείτε. Αυτό θα με χαροποιούσε πάρα πολύ και γιατί είστε γυναίκα. Όλοι λέμε ότι ε, θα πρέπει να στηρίζονται οι γυναίκες. Νομίζω ότι η ΦΑΟ θα βελτιώσει την εικόνα της αν τελικά έχει μια γενική διευθύντρια στους κόλπους της. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ανδρία. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε και, ράς, κυρία Αγγέλα Λανέλ που ήρθατε σήμερα εδώ. Και φυσικά πολύ Γάλλοι ζήτησαν το λόγο, γιατί είχαμε επανειλημμένως ε, και σε πολλά επίπεδα επαφές με την κυρία Αγγέλα Λανέλ. Και είμαστε μάρτυρες ε, της πολύ χρήσιμης συνεισφοράς σας ε, και στην ΕΦΣΑ και στη συνεργασία με την Επιτροπή. Και φυσικά όλοι αυτοί οι παράμετροι συνδυάζονται και με την ε, επιστηστική κυριαρχία και το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων. Πάντως είπατε στην ομιλία σας ε, ότι σας ενδιαφέρουν και τα δύο θέματα και η επιστηστική ασφάλεια αλλά και η επιστηστική κυριαρχία. Και από τη συνεργασία μας καταλάβαμε πόσο αφοσιωμένοι είστε και προσιλωμένοι στα θέματα αυτά και από το πέρασμά σας ε, στο Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας είδαμε πόσο σας ενδιαφέρει και η αγροτική οικολογία. Γιατί πραγματικά ήταν ε, υποδειγματική η παρουσία σας και το πέρασμά σας στο Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας. Σας ε, ενδιαφέρει το θέμα της καταπολέμησης της, ε, του λοιμού στον κόσμο. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια συνάνθρωποι μας υποσυτίζονται, ενώ ταυτόχρονα ένας μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Όλες αυτές είναι σημαντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο ΦΑΟ ε, για τη γεωργία και τα τρόφιμα παγκοσμίω. Χαίρομαι που αυτά τα θέματα είναι προσφυλή ε, και όπως είπατε υπάρχει άρρητος δεσμός μεταξύ της γεωργίας, ε, της διατροφής και της υγείας. Και σίγουρα η ύπεθρος είναι μια δυναμική πραγματικότητα, ένα ζωντανό οργανισμός και χαίρομαι που το αναδείξατε και στην ε, ομιλία σας και ο ρόλος σας θα είναι ζωτική σημασίας για να ξανακατακτήσουμε το χαμένο έδαφος στο όνομα μιας ψευδοβιομηχανοποίησης της γεωργίας που αλλίωσε αυτό τον ε, δεσμό που κανονικά υπήρχε μεταξύ ε, γεωργίας, διατροφής και υγείας. Επίσης, ποια είναι η γνώμη σας για τις ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Γιατί πολλοί προτιμούν να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη και να φέρουμε την προσφορά της γεωργίας στο κοινωνικό σύνολο, στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Πιστεύω ότι μπορούμε να σε έχουμε εμπιστοσύνη γιατί θα προσπίσετε τις αρχές που υποστηρίζουμε και εμείς για τη γεωργία και τη διατροφή. Και χαίρομαι που και το Συμβούλιο σας στηρίζει γιατί δείξατε με τη σταδιοδρομία σας πως ανέκαθεν ακολουθούσατε αυτό το μύτο της Αριάδνης που συνδέει τη γεωργία με τη διατροφή και την υγεία και χαίρομαι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μισελ Νταντάν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε την κυρία Γκέλε Λανέλ για την ομιλία της. Καλώς ήρθατε ή μάλιστα καλώς επιστρέψατε ουσιαστικά στους κόλπους εδώ της ε, Επιτροπής Γεωργίας για αυτή τη συζήτηση και την κοινή αυτή συνεδρίαση με την ΤΕΒΕ. Μιλήσαμε για την επιστηστική ασφάλεια. Εγώ θα δω τα θέματα από κάπω διαφορετική σκοπιά και πρίσμα. Στη διάρκεια τη κοινοβουλευτική ε, θητεία διαπιστώσαμε πόσο ανήμπορη ήταν ε, η Ευρώπη να αντιμετωπίσει μόνη τη την τεράστια αστάθεια των ε, τιμών των τροφίμων παγκοσμίω. Οι διακοιμάσεις ήταν μεγάλες και μάλιστα στην πρόσφατη συναντήση των G20 οι αρχοί κρατών και κυβερνήσεων των πιο πλούσιων χωρών ανέθεσαν μία αποστολή στο ΦΑΟ μία αποστολή παρατήρησης και διαφάνειας. Γιατί γνωρίζουμε ότι η πορεία των τιμών, η εξέλιξη στις τιμές μερικές φορές οφείλεται και σε ψυχολογικούς παράγοντες και στη, στον έλεγχο κάποιων δεδομένων. Ε, γι' αυτό και ήταν απαραίτητη αυτή η αποκατάσταση της διαφάνειας. Τελικά αυτή η αποστολή κάπως χάθηκε ή πέρασε παρατήρητη, κανείς ε, δεν τη σχολιάζει πια ε, ίσως επειδή δεν είχαμε τόσο δραστικές πια διακοιμάσεις στις τιμές ώστε να θεωρηθεί η κοινή γνώμη. Αλλά εσείς τι γνώμη έχετε για αυτό το σκέλος ε, και αυτή την αποστολή του ΦΑΕΟ και πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να ε, υλοποιηθεί αυτή η αποστολή. Δυστυχώς ε, στις 6 πρέπει να μεταβώ σε κάποιες διαπραγματεύσεις αλλά σας διαβεβαιώ ότι ο βοηθός μου θα με ενημερώσει και θα μου διαβάσει τις απαντήσεις σας. Ο κύριος Χόισλινγκ. Ja, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλοι μαζί ευχόμαστε να τα καταφέρετε. Ε, θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Αναφερθήκατε σε κάποια προβλήματα, όμως η πολιτική των ε, τελευταίων ετών ήταν λιγάκι επίμαχη, ε, γιατί ελέγχθησαν πάρα πολλά πράγματα. Ε, νομίζω όμως ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε. Ε, στις δυτικές χώρες το 70% των σιτηρών διοχετεύεται στις ζωοτροφές. Με αυτές τις ζωοτροφές γίνεται πάχυνση και μετά αυτό όμως δεν είναι καλή προοπτική για το μέλλον. Εσείς την όλη συζήτηση πώς τη φαντάζεστε. Από τη μια πλευρά έχουμε εκείνου ε, που θέλουν να προάγουν ε, την βιομηχανοποιημένη γεωργία. Λένε αυτή είναι η λύση, ε, πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλαγμένα προϊόντα. Αλλά αυτή είναι μία άποψη. Η άλλη για την οικολογική γεωργία. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό μοντέλο για την εργασία σας και όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση Έχουμε παγκοσμιοποίηση και στον τομέα της γεωργίας και με όλο και μεγαλύτερη ανησυχία βλέπω ότι όλο και λιγότεροι έμποροι μπορούν να επεκταθούν στις παγκόσμιες αγορές και οι μικρές αγορές κατ' ουσίαν σιγά σιγά εξαφανίζονται. Εσείς λοιπόν τι θέλετε να κάνετε, τι προτίθεστε να κάνετε. Ε, μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου λόγω της παγκοσμιοποίησης θα έχουμε λίγες μόνο μεγάλες εταιρείες, αλλά να μπορούν να επιβιώσουν και οι μικροί γεωργοί. Και τώρα η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε την κυρία για την ε, ε, για όλα αυτά που μας είπε. Άκουσαμε πολλά συναισθηματικά για τη γεωργία, για τη βιομηχανική, της μικρής κλίμακας, ε, την ε, βιολογική γεωργία. Υπάρχουν ίσως δύο στρατόπεδα, οι μεν που τη βλέπουν τη βιομηχανική ως κακή και οι άλλοι που την βλέπουν την οικολογική ως την ιερή γελάδα. Εγώ δεν συμφωνώ με καμία από τις δύο απόψεις. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα υπεύθυνο μοντέλο γεωργίας. Εγώ έρχομαι από μια μικρή γεωργική εκμετάλλευση. Είχαμε 7 ε, παιδιά εκεί στην εκμετάλλευση αυτή, άρα δηλαδή αρκετό προσωπικό. Τώρα όμως αυτή η εκμετάλλευση, η γεωργική εκμετάλλευση πλέον έχει μπει στο βιομηχανικό μοντέλο γιατί δεν υπάρχουν χέρια. Εσείς πώς θα μπορέσετε να επανακαλύψετε τον τροχό γιατί λυπάμαι αλλά έτσι εξελίσσεται η κοινωνία. Και δεν είναι αλήθεια ότι ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, που θέλουν, ξεκινάνε μικρές, ε, θέλουν να μεγαλώσουν. Αυτό ισχύει μόνο για αυτούς ε, που θέλουν να παραμείνουν γεωργοί, γιατί δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που εγκαταλείπουν τη γεωργία και αναζητούν άλλες θέσεις απασχόλησης. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένη απάντηση σε όλα αυτά, αλλά εγώ θέλω να ερωτήσω πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στο ιδανικό μοντέλο για τη γεωργία για την Ευρώπη για τον αναπτυσσόμενο κόσμο και πού θα βρούμε εκείνους που θέλουν να πάνε πίσω στην παλιά εποχή στο να έχουμε το άρωτρο που το σέρνουν ε, ζώα. Γιατί Υπάρχουν δυστυχώς πολλοί που δεν θέλουν να εργαστούν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, είτε είναι βιομηχανικές, είτε πολύ μικρές. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας εύχομαι και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που μας ε, κάνετε. Σας ακούσαμε με μεγάλη προσοχή και μας ενδιαφέρουν όλα τα θέματα τα αγροτικά αλλά και τα θέματα που αντιμετωπίζετε με την αποστολή σας και τη μελλοντική αποστολή σας. Σε κάθε περίπτωση τα τελευταία χρόνια σας ε, σκιαγράφησαν με χαρακτήρα ε, ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων και θα ήθελα να σας πω ότι και το θέμα της επιστημικής ασφάλειας και της επιστημικής κυριαρχίας μας απασχολεί ιδιαίτερα και ε, ως επικεφαλής της ΦΑΟ λοιπόν θα ανταποκριθείτε στις προτεραιότητες αυτές. Η έκθεση που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο θα μας επιτρέψει να απαντήσουμε με καλύτερο τρόπο στα ερωτήματα που θέσατε και στα ζητήματα που μας απασχολούν και που έθεσε και ο Ζήμποβε στα πλαίσια του οργανισμού αυτού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ασφάλεια τροφίμων. Αναφέρετε λοιπόν πολλά ζητήματα τα οποία προφανώς και μας ε, αφορούν άμεσα το θέμα των νέων, των επενδύσεων στον τομέα αγροτικό, το θέμα της καινοτομίας. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αφιερώσει το τμήμα των τα κονδυλίων του Ορίζοντα 2 Ευρώπη για τα τέτοια ζητήματα. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να να δώσει απαντήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά τι αναπτυξιακέ ανάγκε ε, και τις πρακτικές, ε, τις πρακτικές και ε, τόσο προκύπτουν από την αλλαγή κλίματος. Θέσατε και το θέμα της υπαίθρου και αυτό με απασχολεί ιδιαίτερα. Θέλουμε δυναμική υπαίθρο για να συνοδεύσει και τις δραστηριότητες των γεωργών. Δεν αναφερθήκατε όμως στα αγροκτήματα αλλά ως μελλοντική διευθύντρια της ΦΑΟ θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου οι γυναίκες είναι εξαιρετικά ενεργές στην Ήπεθρο και στις γεωργικές δραστηριότητε. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι απλή. Πώς θα προωθήσετε και τις γυναίκες λοιπόν στην Ήπεθρο και στη Γεωργία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ κύριε Νίκολσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά λακωνικό, επιγραμματικό. Ευχαριστώ την κυρία Γκελέν για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τη. Αυτό που με ανησύχησε στην τελευταία πιστιστική κρίση είναι οι μεγάλες διακινήσεις τροφίμων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε την κρίση με το αλογίσιο κρέας. Εκεί χρησιμοποιήθηκαν ε, υπολογιστές για να απολυθούν ε, ποσότητες βοηδών μεταξύ των υπολογιστών έγιναν αυτές οι, οι ε, ενέργειες και πολύθηκαν σε μεγάλες αποστάσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση ε, και αν θα μπορούσαμε να την είχαμε αποτρέψει. Πάντως ε, κάποια δίστακτη βάζουν πολλά χρήματα σε τέτοιου είδους ε, συστήματα που κάνουν κατάχρηση της ψηφιακής δυνατότητας αγοραπολισίας. Είχα πάει και στη Βραζιλία και είδα τι διαφορά έχει η δική τους γεωργία με τη δική μας οικογενειακή γεωργία. Δεν έχει καμία σχέση μια με την άλλη. Δεν ε, ε, υπάρχει ίσω πρόβλημα με το βόλιο κρέα. γιατί οι Βραζιλιάνοι θεωρούν ότι είναι ποιοτικό το δικό τους βόλιο με το δικό μας, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να συναγωνιστούμε το δικό τους γεωργικό εκτινοτροφικό μοντέλο. Και εγώ ω νέο ξεκίνησα σε μια κρατική εκμετάλλευση. Τότε είχαμε και βοήθεια από τα μέλη τη οικογένεια, όπω είπε η κυρία Μαγκίνε. Εκεί όλα τα μέλη τη οικογένεια έβαζαν, έβαζαν το χέρι του και βοηθούσαν στι ε, γεωργικέ δουλειέ. Αυτό δεν ε, συμβαίνει όμω πια. Αν είναι κανεί γεωργό στην Ήπεθρο, δεν πρόκειται να βρει τέτοια βοήθεια. Εγώ μόνος μου να... Ε, αλλά τώρα οι Γεωργοί δεν έχουν την, ε, το χρόνο να ασχοληθούν με τέτοια θέματα. Να κάνουν το ξεβοτάνισμα, για παράδειγμα. Δεν, τα, θέλω να τα βλέπουμε αυτά με ροζ γυαλιά, να τα ωρεοποιούμε, να τα εξοραίζουμε. Η αλήθεια πάντως είναι ότι το παρελθόν έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή και δεν είναι ότι το εξοραίζω, αλλά ό,τι προσπάθηκε να κάνουμε να το επαναφέρουμε έχει παρέλθει. Θα πρέπει όμως οι αγρότες να μπορέσουν να επιβιώσουν στην Ήπεθρο και να έχουμε ένα σύστημα για να στηρίξουμε την, τις αγροτικές κοινότητες και να μπορεί και ο Γεωργός ε, να παράγει τρόφιμα σε τιμές που θα εξασφαλίσουν δική του επιβίωση αλλά και ταυτόχρονα θα είναι σε προσιτές τιμές για τους καταναλωτές. Όλα λοιπόν αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα. Θα μιλήσουμε για τις δασμολογικές ποσοστώσεις, ε, και πώς θα αλλάξει το παλιό σύστημα, αλλά διαρωτώ με προς τα πού οδεύουμε και πώς θα ελέγξουμε όλες αυτές τις εξέλιξεις. Ευχαριστώ και καλή τύχη σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ και αν μου επιτρέπετε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να ε, εκφράσω κάποιες σκέψεις προς την κυρία Αγγελέ που διατέλεσε και εκτελεστική διευθύντρια της του ΕΦΣΑ. Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι μόνο μέρος του προβλήματος, είναι και μέρος της λύσης για την ε, πιστιστική επάρκεια και ασφάλεια. Και μερικές φορές όταν μιλούμε για το διεθνές εμπόριο, είναι σαν να σκεφτόμαστε όπου στέλνοντας εμπορεύματα που περνάνε τον Ατλαντικό κάπου μέσα στον ωκεανό θα γίνει ένα θαύμα και οι τιμές θα πέσουν και θα διατεθούν πιο χαμηλά. Βέβαια όλοι θέλουν να κάνουν εξαγωγές και όλοι ενδιαφέρονται για τις ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Αλλά θα πρέπει να είναι όλοι κερδισμένοι. Και επίσης, μεταφορέ μεταφορές σε τόσο μεγάλες αποστάσεις δεν είναι πάντα απαραίτητε και επηρεάζουν αρνητικά τις κλιματικές αλλαγές. Δύο δισεκατομμύρια, είπατε, συνάνθρωποι μας ε, υποσυτίζονται σε κάποιο βαθμό. Και σίγουρα δεν είναι υπερβολική αυτή η διαπίστωση. και 800 εκατομμύρια να είναι και να μην είναι 2 δισεκατομμύρια που είπατε και πάλι 800 εκατομμύρια είναι υπερβολικός αριθμός για υποσυτισμένα άτομα. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να χορτάσουν την πείνα τους. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, μια επιδημία, μια επιδημία που έχει ξεπεράσει τα περιφερειακά όρια και έχει μετατραπεί σχεδόν σε πανδημία, σε παγκόσμια επιδημία. Και γι' αυτό χρειάζονται και κάποια παγκόσμια μέτρα να αντιμετωπιστεί. Επίσης, ε, ε, ανακύπτουν ε, νέες νόσοι, επιζωτίες ή αρρώστιες των φυτών. Και αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης έχουμε το πρόβλημα της υπερβολικής συγκέντρωσης γεών σε λίγα χέρια. Μερικές φορές ακόμη και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ή χρηματοπιστωτικοί φορείς αγοράζουν μαζικά γεές και κάνουν κατάχρηση της πολιτικής, της γεωρικής πολιτικής, καρπονόμενη κάποιες άμεσες ενισχύσεις. Επίσης, η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και των δύο επιτροπών Άγκρη και Ντέβε συνεργάζονται για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα και γι' αυτό μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε για την μεγάλη συμπάθεια που στο πρόσωπό σας και την αμέριστη υποστήριξη που θα σας προσφέρουμε. Και η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Επιτροπή Ανάπτυξη αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί θέλουμε να αναλυθούν κάποιες παγκόσμιες δράσεις ε, για το διεθνές εμπόριο, όπως είπε και ο επίτροπο ε, ο Φιλ Χόγκαν, αρμόδιο Επίτροπος Γεωργία. Και να μην ξεχνούμε και το πρόβλημα του νερού, γιατί αυτό ταλανίζει ιδιαίτερος τους Γεωργούς. Δεν θα μακρηγορήσω όμως. Θα σας ξαναδώσω το λόγο κυρία Γκελάν για να απαντήσετε στις απορίες των Ευρωβουλευτών και ενδεχομένω να σχολιάσετε αυτά που ακούσατε. Παρακαλώ. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρίες και κύριοι αγαπητοί ευρωβουλευτέ, για την ενθάρρυνσή σα, για την υποστήριξη που εκφράσατε. Είναι σημαντική για μένα. Έχουμε ήδη κάνει σχετικέ εκστρατείε και γι' αυτό λοιπόν εκτιμώ αυτή την ενθάρρυνση και για την τύχη που μου εύχεστε. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσω στις ερωτήσεις σας ε, με τη σειρά. Πολύ αναφερθήκατε. Ο κ κύριος Αντριού στο θέμα της ε, επιστημιστικής κυριαρχίας. Κατανοώ ότι αυτό αποτελεί την δυνατότητα μιας χώρας, την ικανότητα μιας χώρας να αποφασίσει πώς θα τρέφεται ο πληθυσμός της ε, με όλες τις λύσεις που έχει στη διάθεση της, ε, καταρχάς τη δυνατότητα παραγωγής από την ίδια τη χώρα όλων των ε, μερών της διατροφικής αλυσίδας ε, ή τουλάχιστον ενός τμήματος αλλά και προφανώς προς τη θέμενον των ε, στοιχείων των διατροφικών τμήματων που μπορούν να εισαχθούν. Η ΦΑΟ προφανώς θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στις χώρες και στις περιοχές του κόσμου όπου από ό,τι φαίνεται η παραγωγή τροφίμων είναι χαμηλή και είναι ανεπαρκής για να θρέψει τον πληθυσμό. Αλλά και στις χώρες όπου κάποιες χώρες παρέχουν τρόφιμα σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως για παράδειγμα για παράδειγμα, όλες, ε, όλα αυτά τα άτομα τα οποία πάσχουν, που υποφέρουν από υποσυντισμό την υποσαχαρή Αφρική, η Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, στις περιοχές αυτές και στις χώρες αυτές, θα πρέπει να τονώσουμε την αγροτική παραγωγή, η οποία είναι ανεπαρκέστατη και δεν αρκεί να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού δεν είναι μόνο θέμα λοιπόν μόνο της ε, αγροτικής παραγωγής αλλά και της παραγωγής ε, των απαραίτητων τροφίμων και σε ό,τι αφορά την ε, Αφρική στη Ζάμπια για παράδειγμα υπάρχει μεγάλη παραγωγή καλαμποκιού και εξαγωγή του, αλλά ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού εξακολουθεί να πάσχει από υποσυντισμό. Δεν φτάνει λοιπόν να υπάρχει παραγωγή. Πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι τα τρόφιμα που παραγόνται ικανοποιούν τις ανάγκες του πληθυσμού. Νομίζω λοιπόν ότι στον τομέα αυτό θα πρέπει πολλά ακόμα να γίνουν σε πολλές περιοχές του κόσμου. Και προφανώς ε, η ΦΑΟ θα επανέλθω στο θέμα αυτό και θα σας ε, παρουσιάσω τις προτάσεις μου για το πώς θα το πετύχουμε αυτό. Ο κύριος Κολομιέ έθεσε το θέμα της ε, κοινή ε, γεωργικής πολιτικής. Να διευκρινίσουμε ότι η ΦΑΟ συνεργάζεται με όλες τις χώρες του κόσμου για να εξασφαλίσει ότι όλες οι χώρες έχουν την ε, υποστήριξη που χρειάζονται για να αναπτύξουν την σχετική πολιτική στον αγροτικό τομέα και να επιτευχθούν οι στόχοι παραγωγής και βιωσιμότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ίδρυσή της ουσιαστικά από τότε που ίδρυθηκε ως ε, Οικονομική Ένωση αφιερώνει μεγάλη υποστήριξη στον τομέα αυτό και εδώ έχει υπάρξει μεγάλη εξέλιξη όπως γνωρίζετε για να λεφθούν υπόψη και τα οικονομικά στοιχεία αλλά και τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την προστασία του κλίματος, το θέμα της ανάπτυξης της υπαίθρου, προσφάτως και με θέματα κλιματικής αλλαγής. Από την άποψη λοιπόν αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μακρά και πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι πρέπει να αναπραχθεί αυτή η εμπειρία και σε άλλους τομείς, αλλά η βάση περιπτώσει έχει πλούσια εμπειρία. Και πρόσφατα η Παγκόσμια Τράπεζα έκανε μια σχετική έκθεση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και υπολογίζεται ότι 6,5 δισεκατομμύρια παγκοσμίω αφιερώνονται από τις κυβερνήσεις για την υποστήριξη τη γεωργία των χωρών. Και εδώ, αν κοιτάξουμε πώ υλοποιείται αυτή η υποστήριξη, σε κάποιε περιπτώσει έχει να κάνει αυτό με στόχου ω προ την παραγωγή, αλλά και σε ό,τι αφορά στόχους βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας, κλίματος και το καθεξής. Την ε, έκθεση αυτή σας καλώ να την ε, διαβάσετε. Υπάρχει και σύνοψη τεσσάρων σελίδων, γιατί η έκθεση είναι αρκετά μεγάλη. Και εδώ λοιπόν γίνεται μια σύγκριση των σχετικών πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο και παρουσιάζονται και πολύ ενδιαφέρουσες και θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά και την ευρωπαϊκή πολιτική για την υποστήριξη των κοινών αυτών αγαθών. Προστασία του περιβάλλοντος, προστασία από την αλλαγή του κλίματος, ανάπτυξη της υπαίθρου και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ο κόσμος ε, έχει ως προσδοκίες από την γεωργία. Ο κ. Σέρτος αναφέρθηκε στην ασφάλεια των τροφίμων. Έχετε δίκιο. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της ε, επιστημιστικής ασφάλειας. Θα πρέπει να παρέχεται στους πολίτες σωστή και θρεπτική διατροφή σε επαρκείς ποσότητες και σε τιμές ε, προσβάσιμες στον καταναλωτή. Ποιος είναι ο ρόλος της ΦΑΟ στο σημείο αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολυδιάστατος. Να σας αναφέρω και πάλι το γεγονός ότι η ΦΑΟ και η ΠΟΗ μαζί με την Αφρικανική Ένωση πριν από κάποιες ημέρες διοργάνωσαν στην Αντισαμπέμπα μια στην ΑΔΡΙΟ για την ασφάλεια των τροφίμων. Έγιναν πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις προφανώς για το πώς μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη τεχνική αρρωγή προκειμένου να υπάρξει αυτό που ονομάζουμε capacity building, ανάπτυξη δυναμικού στις χώρες για να αυξηθεί το επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας των τροφίμων. Όλος ιδιαίτερος στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αυτό που με έκανε εντύπωση στο συνέδριο αυτό ήταν το εξής το θέμα του εμπορίου και των εξαγωγών δεν ήταν ε, σε κεντρική θέση γιατί θα υπάρξει ένα ειδικό συνέδριο την Άνοιξη για τα θέματα αυτά και ουσιαστικά αυτό που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε ότι το θέμα αυτό της ασφάλειας των τροφίμων αφορά καταρχάς την ε, υγεία των δικών μας ε, πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλες τις χώρες του κόσμου να εξασφαλίσουμε ότι πετυχαίνουμε τα πρότυπα αυτά τα οποία θα μας επιτρέψουν τελικά να προστατεύσουμε τους καταναλωτές μας. Και εδώ διαδραματίζει σημαντικό και κεντρικό ρόλο η ΦΑΟ σε ό,τι αφορά την τυποποίηση, για παράδειγμα, του κόντεξ αλμιμετάριους. Εδώ, σε παγκόσμιο επίπεδο, με όλες τις κυβερνήσεις πρέπει να πετύχουμε πρότυπα τα οποία με τη σειρά τους θα μας επιτρέψουν να συμφωνήσουμε επί των κανόνων που θα πρέπει να ισχύουν και στις ανταλλαγές, καθότι αυτά τα πρότυπα αποτελούν σημαντικά πρότυπα αναφοράς από τον ΠΟΕ, αλλά τα πρότυπα και οι προδιαγραφές αυτές θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι χρησιμοποιούνται και από πολλές αναπτυσσόμενες χώρες εντάσσονται στην νομοθεσία τους για να προστατεύσουν με τη σειρά τους και τους δικούς τους καταναλωτές. Και εδώ λοιπόν η ΦΑΟ θα πρέπει να τονίσει ότι οι προδιαγραφές του Κόντεξ Elementarius δεν έχουν μόνο εφαρμογή στο εμπόριο τροφίμων, προφανώς έχουν και εκεί εφαρμογή, αλλά και ότι αποτελούν και βάση για την προστασία των καταναλωτών, ανεξαρτήτως από τη χώρα στην οποία ζουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά Όσον αφορά την ε, οικολογική γεωργία, αν θυμάμαι καλά αυτός ο όρος χρησιμοποιήθηκε, ο στόχος όπως είπατε και εσείς είναι πρώτα απ' όλα να μειωθούν οι απώλειες, οι ζημιές και οι σπατάλοι Πριν από λίγες εβδομάδες μίλησα σε κάποιους Καναδούς και μου είπαν ότι το 40% των παραγόμενων τροφίμων στον Καναδά ε, σπαταλιούνται, πετιούνται Άρα δηλαδή ε, στην, ε, στο, σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το προσέξουμε αυτό, να μην έχουμε τέτοιου είδους ε, ζημιές. Όταν μιλάμε για την βελτίωση της παραγωγικότητας, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη δυνατότητά μας σε 20, 30, 40 χρόνια να μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε τρόφιμα έτσι ώστε να έχουμε και παράλληλα υγιή, εδάφη, καλή ποιότητα νερού. Άρα δηλαδή η γεωργική οικολογία, μάλλον η γεωργία περισσότερο, είναι μία προσέγγιση που βοηθάει στο να συνδυάσουμε ε, την οικολογική και την οικονομική απόδοση της γεωργίας μας. Ε, δεν είναι βέβαια μία μόνο προσέγγιση, αλλά είναι μία σειρά ε, προσεγγίσεων που μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η οικολογική μορφή της γεωργίας. Αυτό έχει ήδη γίνει τα τελευταία χρόνια, το έχει ήδη πράξει η ΦΑΟ. Κατόπιν αναφερθήκατε στις ε, επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι ο πυρήνας του προγράμματός μου. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτούς τους τομείς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς του παρελθόντος που κατ' ουσίαν αποτελούν το μέλλον μας. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικέ επενδύσεις. Η ΦΑΟ δεν είναι βέβαια επενδυτικός οργανισμός, έχει ένα πρόγραμμα τεχνικής συνεργασίας, αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ ενδιαφέρον ε, και εγώ φιλοδοξώ να το ε, δηλαδή η ΦΑΟ ε, χρηματοδοτεί κάποια προγράμματα. Η ΦΑΟ μπορεί να δείξει ε, ποιες είναι οι επιτυχίες ε, που σημειώνονται για να έχουμε καλύτερη παραγωγή. Εγώ λοιπόν θέλω να εξηγιάνω αυτό το πρόγραμμα. Όμως αυτό το πρόγραμμα παραμένει περιορισμένο με την έννοια ότι έχει περιορισμένη χρηματοδότηση, είναι βραχυπρόθεσμα τα προγράμματα και όπως ε, σας είπα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας αν θέλουμε να μπορούμε να προσφέρουμε τρόφιμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πεινάνε και ποσιτίζονται. Άρα δηλαδή η όλη ιδέα είναι ε, να μπορέσουμε να προβούμε σε μεγαλύτερες επενδύσεις και μέσω της ΦΑΟ. Και αυτό ε, μπορούμε να το κάνουμε με τη στήριξη της ΦΑΟ αλλά και με τη συνεργασία με διώτες ε, και με δημόσιους επενδυτές. Η ΦΑΟ ήδη το κάνει αυτό. Αναφέρθηκα στις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει η ΦΑΟ ε, με την ε, Παγκόσμια Τράπεζα και με την IFAD, ε, τη Διεθνή Τράπεζα Γεωργικής Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκεί η ΦΑΟ προσφέρει τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη σε αυτούς τους οργανισμούς για να μπορούν να εφαρμόσουν συγκεκριμένα επενδυτικά προγράμματα. Μιλάμε σήμερα για 5 δις δολάρια επενδύσεων που δεν είναι άσχημα αλλά δεν αρκούν κατά την άποψή μου. Άρα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες του οργανισμού. Ε, μπορεί να γίνουν όλα αυτά σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά και με πολλούς άλλους ε, χρηματοδότες. Έχω κατά νου κυρίως ε, περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες, τις οποίες μπορεί να στηρίξει η ΦΑΟ. Όπως σας είπα, πρέπει να αναπτύξουμε την αλυσίδα αξίας στις γεωργικές περιοχές για να διασφαλίσουμε αυτό που λέει και η Παγκόσμια Τράπεζα, ότι η γεωργία και η αλία είναι οι τομείς που είναι οι πιο αποτελεσματικές αποτελεσματικοί μπορούν να προσφέρουν στο να αντιμετωπιστεί η πείνα. Οι περισσότεροι φτωχοί στον κόσμο ζουν σε ε, γεωργικές ε, περιοχές και οι περισσότεροι από τους φτωχούς είναι γεωργοί και αλείς. Γι' αυτό λοιπόν ε, αν αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα θα είμαστε αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση της πείνας. Πρέπει σε αγροτικές περιοχές να αναπτύξουμε οικονομικές δραστηριότητες με επίκεντρο την γεωργία και την αλεία. Έχω κατά την μεταποίηση τροφίμων, συσκευασία, τη χιλιανική πώληση τροφίμων. Όλες αυτές τις δραστηριότητες πρέπει να τις αναπτύξουμε σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές. Και όλα αυτά συμβαίνουν κυρίως στην Ασία. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τη σχέση ανάμεσα στη ΦΑΟ και αυτούς τους επενδυτές, όχι ε, με την έννοια ότι η ΦΑΟ θα είναι επενδυτής, αλλά η ΦΑΟ θα δώσει σε όλους αυτούς τους επενδυτές τη γνώση ε, και την τεχνογνωσία που διαθέτει, έτσι ώστε να εφαρμοστούν επενδυτικά προγράμματα στις γεωργικές περιοχές. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, να παραμείνουν οι νέοι στη γεωργία και να μην μπαίνουν σε πειρασμό ή να μην εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις γεωργικές περιοχές για να πάνε σε μια άλλη πόλη ή σε άλλη ε, χώρα ή σε άλλη πυρο. Αυτός είναι ο στόχος μου. κατόπιν. Κύριε Χαγκούσκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αναφερθήκατε στις γυναίκες. Πράγματι, ε, στην ομιλία μου δεν αναφέρθηκα στις γυναίκες, ε, παρότι οι γυναίκες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα επισητιστικά συστήματα. Βρισκόμαστε τώρα παντού. Οι γυναίκες βρίσκονται στα χωράφια, βρίσκονται στα εργοστάσια που μεταποιούν τρόφιμα, βρίσκονται στα καταστήματα, βρίσκονται παντού. Οι γυναίκες ε, δεν ε, αναγνωρίζεται πάντα η προσφορά τους, ούτε ο ρόλος τους ε, στα επιστημιστικά συστήματα ε, και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια, έχουν μερικές φορές δυσκολία στο να αποκτήσουν πρόσβαση σε γη. Έχουν δυσκολία να αποκτήσουν πρόσβαση σε φυσικούς πόρους. Και οι γυναίκες επίσης πολλές φορές δεν συμμετέχουν ε, στο επίπεδο που λαμβάνονται αποφάσεις για τη γεωργία, για την αλία. Άρα δηλαδή οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι όποια ενέργεια και αν αναπτύξει η ΦΑΟ οφείλουμε να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο να ε, καταρτιστούν κριτήρια επιλογής έτσι ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα, να βελτιωθούν οι δυνατότητες των γυναικών. Θα το προσέξω πάρα πολύ αυτό, γιατί νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε θετική επίδραση στο επισητιστικό σύστημα και στην ασφάλεια των τροφίμων. Αναφερθήκατε και στην Κοινοβουλευτική Συμμαχία κατά της φτώχειας. Συγχαρητήρια. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική αυτή η πρωτοβουλία. Δική μου φιλοδοξία είναι να ξαναβάλουμε τη γεωργία, την, την αλληλεία, την ασφάλεια των τροφίμων ως ύψιστη προτεραιότητα το πολιτικό μας προγράμματο και σίγουρα αυτό συμβαδίζει και με τη δική σας πρωτοβουλία. Και μακάρι και τα Εθνικά Κοινοβούλια να προσχωρήσουν σε αυτή την πρωτοβουλία, όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη αυτή η πρωτοβουλία και αν εκλεγώ πραγματικά διοριστώ θα... Ε, συμβάλλω και εγώ σε αυτή τη δική σας την κοινοβουλευτική προσπάθεια κατά πολέμηση της φτώχειας στον κόσμο. Έχω πολλά ακόμη να πω, αλλά διαπιστώνω ότι μας έχει μείνει ελάχιστος χρόνος. Θα ήθελα πάντως να απαντήσω στην ερώτηση που μου έκανε κάποιος για το τι γεωργικό μοντέλο ε, υπερασπίζομαι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά γεωργικά μοντέλα στον κόσμο. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι Παγκοσμίω η γεωργία μικρής κλίμακας είναι αυτή που εξασφαλίζει την μεγαλύτερη ασφάλεια των τροφίμων και η μικρή εμβέλεια γεωργία συμβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό στην παγκόσμια επιστηστική ασφάλεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη, σίγουρα η κατάσταση εκεί διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα και σίγουρα στη... στην Αφρική έχουμε μεγάλα ευρύτατα γεωργικά συστήματα ε, για να αντιμετωπιστούν οι στόχοι της επιστηστικής ασφάλειας ε, που έχει χώρα αυτή η Νότια Αφρική, παράδειγμα. Η Βραζιλία, όντως, ε, εκεί υπάρχουν τεράστιες φάρμες, αλλά η ασφάλεια τροφίμων της χώρας αυτής βασίζεται κυρίως στην γεωργία μικρής κλίμακας, όχι στις απέραντες εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις. Οπότε υπάρχουν διάφορα γεωργικά μοντέλα. Το θέμα είναι το μοντέλο που θεωθετήσουμε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε γεωργού και να μπορεί εν ανάγκη να αυξήσει την παραγωγικότητά του. Και εδώ σκέφτομαι κυρίως αυτούς τους μικροκαλλιεργητές που θέλουν να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους και θέλουν να αναπτύξουν μια πιο επικερδή δραστηριότητα, ώστε να μην ε, καταφέρουν απλώς να βιοποριστούν και να επιβιώνουν, αλλά να μεταβούν σε μια πιο εμπορική γεωργική δραστηριότητα, πιο κερδοφόρα. Βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει με βιώσιμο τρόπο. Και επίσης και οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις να είναι βιώσιμες, γιατί και αυτές θα πρέπει να μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε τους φυσικούς μας πόρους και να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Και υπάρχει κάτι που Όλοι έχουμε ως κοινό στοιχείο, άσχετα με το οργικό μοντέλο που έχουμε επιλέξει, το θέμα της γύρεσης του πληθυσμού, το δημογραφικό πρόβλημα που παρατηρούμε παντού στον κόσμο. Οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε να προσεγγίσουμε περισσότερους νέους στη γεωργία για να εξασφαλίσουμε αυτή την ηλικιακή ανανέωση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλίας στον κόσμο. Και ένα τελευταίο σημείο για την παγκοσμιοποίηση αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στην ερώτησή σας για την παγκοσμιοποίηση. Ρωτήσατε αν η παγκοσμιοποίηση είναι πρόβλημα ή λύση. Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα γεγονός. Είναι γεγονός η παγκοσμιοποίηση και φυσικά δεν σας λέω τίποτα καινούριο. Όλοι το γνωρίζουμε και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε από τους πρώτους εισαγωγής και εξαγωγής παγκοσμίω σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η παγκοσμιοποίηση αυτή να γίνεται σε δίκαιες βάσεις, να προστατεύει τους πιο αδύναμους και κυρίως τις χώρες που σας ανέφερα, τις φτωχότερες χώρες, και εκεί που διαμένουν οι φτωχότεροι γεωργοί κτηνοτρόφοι και αλείς. Και φυσικά υπάρχει το θέμα της ρύθμισης της παγκοσμιοποίησης. Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε την παγκοσμιοποίηση με πολυμερή συστήματα όπως τη Παγκόσμια Οργάνωσης Εμπορίου και μάλιστα θα μεταβούμε στη Γενέβη για να συναντήσουμε εκπροσώπους ΠΟΕ και να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να λάβουμε υπόψη και το πρόβλημα που έχουν οι φτωχότεροι και οι πιο εκτεθειμένοι στι μεγάλε διακοιμάνσει των τιμών, αλλά και στη συνέπεια των κλιματικών αλλαγών. Αυτοί χρήζουν προστασία. Είναι πιο αδύναμοι. Θα πρέπει λοιπόν να του βοηθήσουμε να εξασφαλίσουν την επιβίωσή του και την επιστηστική του ασφάλεια. Και ο ρόλο του κόντεξ αλιμεντάριο είναι πολύ σημαντικό. Ώστε αυτή η παγκοσμιοποίηση να είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει σε βάση που θα προστατεύουν τον καταναλωτή, την υγεία του, αλλά και την ενημέρωσή του, ώστε εμπεριστατωμένα να μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Αυτές, ε, κύριε Πρόεδρε, είναι οι απόψεις μου για την παγκοσμιοποίηση. Σίγουρα πάντως ε, αυτό το θέμα βρίσκεται στο επίκεντρο της εντολής ε, του Γενικού Διευθυντή του ΦΑΟ και σίγουρα θα συνεργαστώ με τους αρμόδιους φορείς για τα θέματα αυτά. Και τέλος, και εδώ θα ολοκληρώσω, με την τελευταία σας ερώτηση για το τι θα πρέπει να κάνουμε και πώς θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε όλους αυτούς τους στόχους, να καταπολεμήσουμε τις επιζωτίες, τις αρρώστιες των φυτών, να καταπολεμήσουμε την πείνα και τον υποσυτισμό, ε, την αρπαγή των γεών την υπερβολική συγκέντρωση των γεών, την παχυσαρκία και το καθεξής. Σίγουρα χρειάζονται γνώσεις, χρειάζεται εμπειρογνωμοσύνη, χρειάζεται στοχευμένη ανάλυση, αλλά θα πρέπει αυτή τη, αυτή τη γνώση, αυτή την εμπειρογνωμοσύνη και την ανάλυση να την ε, μετατρέψουμε σε δράση. Και γι' αυτό η προτυποποίηση, ε, η ρύθμιση και οι εθελοντικές κατευθυντήρες γραμμές ε, να διέπουν τις υπεύθυνες επενδύσεις ώστε να περιορίσουμε αυτή τη συγκέντρωση των γεών, την αρπαγή των γεών που είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο. Έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ε, στις ανησυχίες ε, και τα προβλήματα που αναφέρατε. Αυτά λυπούμε λοιπόν, που δεν μπόρεσα να επεκταθώ περισσότερο, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ νομιωτική αυτή συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και του συναδέλφους για τις πολύ καλές και εύστοχε ερωτήσει που έθεσαν. Η συνεδρίαση αυτή καταδεικνύει πόσο χρειαζόμαστε στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε κοινέ προσπάθειες για να πετύχουμε την εκρίζωση της φτώχειας και της πείνας μέχρι το 2030. Ειλικρινά ελπίζω ότι η συνεργασία με τη Μελλοντική Γενική Διευθυντρία της ΦΑΟ θα είναι και ένα κίνητρο στις ε, επερχόμενες ευρωεκλογέ. Σε ό,τι αφορά θέματα απασχόλησης, επιστικής ασφάλειας, ε, και κρίζωσης ε, του λοιμού στις ε, αφρικανικές χώρες αλλά και στις υπόλοιπες χώρες. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί οι, τα παραδοσιακά εργαλεία θα πρέπει να ανανεωθούν. Χρειαζόμαστε νέα εργαλεία και ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη λοιπόν συνεργασία και καλύτερο συντονισμό σα. Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία για την εκλογή σα και θα παρακολουθήσουμε τη διαδικασία με μεγάλη προσοχή. Σα ευχαριστώ όλου. Μάλιστα, να σας υπενθυμίσω αγαπητοί συνάδελφοι ότι αύριο Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι αύριο 9 με 11 θα συνεδριάσουν οι συντονιστέ και κατόπιν θα έχουμε την δημόσια συνεδρίαση τη Επιτροπή Γεωργία. Σα ευχαριστώ. Καλό σα βράδυ.